Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Οντή, βεβαίω είναι θέμα επί του κανονισμού, είναι θέμα σχετικό, θα επιληφθούμε και κατατίθενται τα πρακτικά στην έναρξη της προσοχής συνόδου, εάν δεν εκφραστούν αντιρρήσεις, εγκρινούνται και τα σχετικά ψηφίσματα, εάν δεν υπάρξουν αντιρρήσεις στα αρμόδια όργανα, αντιρρήσεις δεν